Έχουμε την παρουσίαση της εκθέσεως Καμπεζόν Ρούις για τις δραστηριότητες ε, του διαμεσολαβητή για το 2014. Θέλω να καλωσορίσω και την κυρία Ρέιλι, την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Η κυρία Καμπεζόν Ρούις έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ε, κύριε Επίτροπε. Το Ευρωβαρόμετρο λέει ότι το 40% των Ευρωπαίων πολιτών έχει εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά όργανα. Ο διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής προσπαθεί να βελτιώσει ε, την, σε επιδόσεις αυτές ε, και στα πλαίσια της αύξησης της ε, διαφάνειας ερευνά ο διαμεσολαβητής ε, ε, τις διάφορες περιπτώσεις ε, όπου πιθανολογείται αρνητική μορφή διαχείρισης των ευρωπαϊκών υποθέσεων και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ρέιλι και την υπηρεσία της τον καιρό που είναι υπεύθυνη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά αντιμετωπίζει με, έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα πάνω από 2.325 υποθέσεις. Θα ήθελα να πω ότι έχει πάρα πολύ σημασία ε, ότι έχει ασχοληθεί και με θέματα μείζωνος σημασίας για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό και στρατηγικής ε, σημασίας για ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει σαν παράδειγμα μια πολύ μεγάλη όθηση στις προσπάθειες για βελτίωση της διαφάνειας στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων TTIP. Έχει επίσης ε, προωθήσει τα θέματα διαφάνειας για την παρουσία των ομάδων συμφερόντων ιδιαίτερα στα πλαίσια της επεξεργασίας της, του νέου κανονισμού της κοινή αγροτικής πολιτικής που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ε, Έχει πολλές παρεμβάσεις και στα θέματα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως επίσης και στο θέμα της δυνατότητας των προσφύγων να κάνουν ε, προσωπικές ε, αναφορές για θέματα τα οποία τους αφορούν. Δεν θα πρέπει να χάσουμε λοιπόν την ευκαιρία ε, για να πούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει την τεράστια αυτή προσπάθεια η διαμεσολαβήτρια και να υπογραμμίσουμε επίσης πόσο μεγάλη σημασία έχει για τους πολίτες ιδιαίτερα στην σε τομεί όπως η προστασία των καταναλωτών, η προστασία της υγείας και η προστασία των εργαζομένων. Πρέπει να συνεχίσει να αναζητεί εγγυήσει στα πλαίσια των σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στα πλαίσια της σοβούσης προσφυγικής κρίσης εδώ οδηγίες όπως η επικύρωση της συνθήκης ε, του Μαρακέσα ή ε, η επεξεργασία της νέας οδηγίας είναι θέματα τα οποία, ε, στα οποία η παρέμβαση της διαμεσολαβήτριας είναι σημαντική. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να πω ότι αναγνωρίζουμε την τεράστια προσπάθεια την οποία έχει κάνει η υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περίοδου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών για το εξαιρετικό κλίμα εργασίας και γι' αυτό μπορέσαμε να καταλήξουμε σχετικά γρήγορα στην παρούσα πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Καμπεσόν. Έχει το λόγο τώρα η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Να ευχαριστήσω την ε, κυρία Καμπεθόν Ρουίθ αλλά και όλους τους κοιόδες ηγητές ε, που εργάστηκαν τους τελευταίους μήνες για αυτήν την έκθεση. Με το κείμενο αυτό βλέπω ότι κατανοείτε και στηρίζετε τη στρατηγική μου για το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Έχω πει επανειλημμένως ότι δεν θα μπορέσω να ασκήσω το λειτουργήμά μου όπως πρέπει χωρίς ε, την υποστήριξη του κοινοβουλίου την οποία έχω λάβει τόσο εγώ όσο και η προκάτοχή μου μέχρι τώρα. Είμαστε ένα μικρό γραφείο, λιγότερο από 80 μέλη προσωπικού, όμως έχουμε μια μεγάλη αποστολή για τους πολίτες της Ευρώπης και θα προσπαθήσω να διαδραματίσω το ρόλο μου βοηθώντας τα θεσμικό όργανα της Ένωσης ε, να ε, μη αρθούν στο ύψος των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών. Κυρίως δε μετά από τα γεγονότα των τελευταίων ε, ημερών, μηνών, ετών. Σας ευχαριστώ για αυτή την υποστήριξη. Έχουμε συμπληρωματικούς ρόλους. Εργαζόμαστε όχι εν κενό, αλλά άμεσα σε συνεργασία με τους πολίτες, γιατί αυτοί έρχονται ζητώντας βοήθεια ή για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε εμάς. Ιδίω όταν είπε ε, και ο αντιπρόεδρος Τίμερ μας και το έχει πει πολλές φορές, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία θα πρέπει να υποστηριχθούν ε, και να απορασπιστούν ακόμη πιο έντονα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για δεύτερη φορά έρχομαι στην Ολομέλεια. Είχα έρθει και τον Οκτώβριο, πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2013. Έχω έρθει και σε επιτροπές του Κοινοβουλίου, Επιτροπή Αναφορών, Ελέγχου του Προπολογισμού, Απασχόλησης, Νομικών Υποθέσεων, Πολιτικών Ελευθεριών και κάθε φορά έχω επωφεληθεί τα μάλα από την εμπειρία, τη στήριξη και αυτό πιστεύω ότι φαίνεται και σε στρατηγική που έχω αναπτύξει και εφαρμόζω. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών που ε, επικρότησε την στρατηγική μου για τον προτέρων έρευνες. Χρησιμοποίησα αυτή την στρατηγική προσέγγιση για να ξεκινήσω το διάλογο στο ανώτατο δυνατό επίπεδο για να βοηθήσω τους διάφορους θεσμούς ε, να πετύχουν τα ανώτατα πρότυπα δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, το γραφείο μου είναι και πάντοτε ε, θα είναι ο κόμβος υποδοχής ε, καταγγελιών. Το 20% των καταγγελιών σήμερα ε, έχουν να κάνουν ε, με άρνηση σε πρόσβαση σε έγγραφα. Η διαφάνεια, το δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα που κατοχυρώνεται από τη συνθήκη πρέπει να ε, κατοχυρώνεται γιατί είναι θέμα δημοκρατικής συμμετοχής και δημοκρατικής λογοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά καθορίζει ανώτατα όρια και πρότυπε, ω ανώτερα από άλλων κρατών αλλά ε, θα πρέπει ε, να προσπαθεί να τα ε, αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καμπεθόν Ρουίθ που στηρίζει την προσέγγιση μου σε ό,τι αφορά το λεγόμενο, τις λεγόμενες περιστρεφόμενες πόρτες, δηλαδή την αλλαγή καθηκόντων κάποιων δημόσιων λειτουργών που αναλαμβάνουν μετά ένα πολιτικό αξίωμα. Είναι θετικές οι εξελίξεις αυτές και για πρώτη φορά βλέπουμε ότι η Κομισιόν δημοσιεύει τον κατάλογο ε, των ανώτερων υπαλλήλων ε, που έφυγαν και πήγαν ε, σε άλλες θέσεις και ενδέχεται να υπάρχει εκεί κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Με βάση τον υπηρεσιακό κανονισμό θα δημοσιεύεται ετησίως ο κατάλογος αυτός και η Επιτροπή Περιπολισμού έδωσε τη δέουσα σημασία στο σημείο αυτό. Αναγνωρίζει επίση η έκθεση την πραγματική πρόοδο που σημείωσε η Κομισιόν μετά από δική μου έρευνα και πίεση και από το Κοινοβούλιο για τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων τη συμφωνία TTIP. Αυτό ήταν κατ' εξαιρετικό παράδειγμα τη συνεργασία Κοινοβουλίου, Επιτροπή και Διοικήσεων. Το θέμα επίσης ε, της διαφάνειας ε, των ομάδων πίεσης, του lobbying, ήταν κάτι σημαντικό. Ε, υπάρχει μια πρωτοβουλία διαφάνειας, στην ενθαρρύνω και βλέπω ότι γίνεται ήδη μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο κομισιών. Σε ό,τι αφορά την καπνοβιομηχανία, έχουμε ένα ζήτημα, θα συζητηθεί σύντομα στο Κοινοβούλιο. Πρόσφατα έλαβε η Κομισιόν απόφαση να μην δεχτεί τη σύστασή μου για την εκ των προτέρων δημοσιοποίηση των συναντήσεων με τον κλάδο αυτό. Λυπούμε γι' αυτό η, ε, το νομικό δεσμευτικό πλαίσιο, η σύμβαση για τον έλεγχο του καπνού των ΗΠΑ ε, την έχει προσυπογράψει η Ένωση, αναγνωρίζει ε, την ε, καπνοβιομηχανία ως έναν από τους παρούς, ο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι συνήθεις διατάξεις ε, σε ό,τι αφορά το διάλογο. Επίσης, ε, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δημοσιοποιεί πλέον ε, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του. Ο Μάριο Ντράγκη συνεργάστηκε μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό για την δημόσια εμπιστοσύνη και τον ευχαριστώ. Επίσης, θέλω να δω και τι θα πει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά την έρευνά μου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις ομάδες πολιτικού διαλόγου στα θέματα γεωργίας. Δημόσιες διαβουλεύσεις για τη βελτίωση του Μητρώου Διαφάνειας είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί ε, με ένα τέτοιο Μητρό θα μπορούμε να έχουμε την πλήρη διαφάνεια. Όλοι να ξέρουν ακριβώς ποιο και πού έχει καταχωρηθεί και αν έχει και πού πρόσβαση για τη διαδικασία λήψεων αποφάσεων. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια για τι κλινικέ δοκιμέ, το ανέφερε η κυρία Καμπεθόν, ξέρω ότι την ενδιαφέρει, ε, θα συνεχίσω την έρευνα σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων των κλινικών ε, δοκιμών, σε ό,τι αφορά ένα πάρα πολύ ακριβό φάρμακο, το χουμίρα, δις κόστησε. και θέλω να δω επίσης τι γίνεται και στα θέματα μετανάστευση και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω του βουλευτέ για τη μεγάλη του υποστήριξη ε, στην ειδική έκθεση του, που έκανα στο Κοινοβούλιο ε, σε ό,τι αφορά την άνιση του Frontex να ε, καθιδρύσει ένα μηχανισμό επίλυση διαφορών. το Κοινοβούλιο όμω δέχθηκε τι συστάσει μου για αυτό το μηχανισμό και για τη μεταχείριση των ατόμων που απελάβνονται από, την Ένωση δυνάμει των προτάσεων του Frontex. Επίσης έχω εργαστεί στον τομέα των καταγγελών των θεμελιωδόμων δικαιωμάτων, πολιτικής συνοχής, χαιρετής τις προσπαθειές μου η κυρία Καμπεθών. Επίσης δικαίωμα τα ανθρώπων με αναπηρία Σε σχετική σύμβαση, επίση έχουμε κάνει δουλειά. Ε, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συγγόνο του Πολίτη, προεδρεύω αυτού του δικτύου, κάνουμε παράλληλες έρευνε σε θέματα που αφορούν Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικά οριζόντια επίπεδα. Είναι ένα νέο εργαλείο αυτό ε, και θα γίνει στις Βρυξέλλες ε, μια διάσκεψη του δικτύου. Όλοι οι Εθνικοί Περιφερειακοί Σύνηγοροι του Πολίτη θα έλθουν για να συζητήσουμε ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Και αυτό δεν θα είναι μια ευκαιρία μόνο σε εμά σε επίπεδο Ένωσης να διδαχθούμε από τις εμπειρίες των συνηγόρων του πολίτη, αλλά και αυτοί θα διδαχθούν από το τι κάνουμε εμείς καλά εδώ στα θεσμικά όργανα και πολλές φορές αυτά περνούν απαρατήρητα. Και θα σας αποστείλω την πρόσκληση σύντομα για αυτό το συνέδριο, αυτή τη διάσκεψη. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τις ε, καταγγελίες, είχαμε ένα αριθμό 80%. Ξέρω ότι υπάρχει αυτό το ποσοστό 20% μη συμμόρφωσης ε, το είδατε στην ετήσια έκθεση του 2014. Ήδη μπορώ να σας πω από τώρα όμως ότι για το 2015 στην ετήσια έκθεση έχουμε 90% ποσοστό συμμόρφωσης. Πολύ ικανοποιητικό επίτευγμα. Δεν θα ήταν δυνατόν εάν δεν είχαμε την αυξανόμενη υποστήριξη όλων των οργανισμών, όλων των θεσμικών οργάνων και βέβαια πιο πολύ του Κοινοβουλίου. Πριν ολοκληρώσω να πω ότι πρέπει να καταγραφεί για μια ακόμη φορά το πόσο με έχουν εντυπωσιάσει τα πολύ ψηλά πρότυπα ε, των δημόσιων υπηρεσιών, των χιλιάδων αυτών υπαλλήλων της Ένωση ε, των οργανισμών, θεσμικών οργάνων. Οι περισσότεροι από αυτούς ε, δουλεύουν σκληρά, ε, δείχνοντας επαγγελματισμό ηθική. Υπάρχει επίσης ανανέωση της αξιοπιστίας της κοινή γνώμης απέναντι στους θεσμούς και έχουμε αυτή την πολιτική πρόκληση να εξασφαλίσουμε την ηθική υπεύθυνη δημόσια δίκηση που ενδυναμώνει τη δημοκρατία. Για να πετύχουμε υψηλότερα επίπεδα νομιμοποίησης θα πρέπει σε επίπεδο δημόσιας δίκαιη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ποιότητα αλλά και να στηρίζουμε στόχους, διαφάνεια, ηθική, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα. Ω Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια θα εργαστώ με τα θεσμικά όργανα, με του εκτελεστικού οργανισμούς, με το κοινοβούλιο σα ε, για να πετύχουμε αυτού ε, τους στόχους. Ολοκληρώνοντα, θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την εισηγήτρια, τους σκιώδει εισηγητέ, το προσωπικό, τη γραμματεία για όλη σε τη δουλειά και περιμένω να ακούσω με ανυπομονησία τις δικές σας παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Ms. Ευχαριστώ κύριε Ορέλη. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο Τίμερμαν. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Καμπεθόν Ρούις, για την εξαιρετική ε, παρουσίαση για τις εργασίες της διαμεσολαβήτριας το 2014. Η καταπολέμηση των καταχρηστικών μορφών διοίκησης και διαχείρισης είναι ο κοινό μας στόχος. Και γι' αυτό ακριβώς και η ισπανική μετάφραση της λέξης διαμεσολαβητής ombudsman περιγράφει με σωστό τρόπο την λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, defensor de pueblo, υπερασπιστής του λαού. Ε, θέλω επίσης να σημειώσω την συστηματικά καλή συνεργασία με την ε, κυρία Ρέιλι και τις υπηρεσίες της. Θα σχολιάσω τη σημασία των εργασιών της διαμεσολαβήτριας στον τομέα της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους στον τομέα της διαφάνειας και αυτό αναγνωρίζεται στην έκθεση Καμπεσον από την 1η Δεκεμβρίου του 2014 ε, στους επιτρόπους, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές των γραφείων πρέπει να ε, καταθέτουν ένα κατάλογο ε, με τις ομάδες συμφερόντων με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή απαιτήθηκε επίσης υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων TTIP και εδώ είχαμε και πολύ έντονες ε, ανταλλαγές επιχειρημάτων και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαμεσολαβήτρια υπογράμμισε την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ θέλω να συγχαρώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βοήθησε προς την κατεύθυνση αυτή. Η πλειοψηφία των συστάσεων του Ombudsman της διαμεσολαβήτριας μάλλον σχετικά με τις περιστριφόμενες θύρες, δηλαδή τις ανταλλαγές θέσεων των ανωτέρων υπαλλήλων, όπως επίσης και την λειτουργία τους μετά από την αποχώρησή τους, αμέσως μετά από την αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί τομείς όπου οι συστάσεις της διαμεσολαβήτρια ακολουθήθηκαν από πλευράς μας. Πήραμε τα μέτρα έτσι ώστε η πρωτοβουλία των πολιτών να γίνει πιο χρηστική, προς, πιο φιλική μάλλον προς τους χρήστες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει επίσης και έναν μηχανισμό παραπώνων για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της διαμεσολαβήτριας στα πλαίσια της έρευνας για το Frontex. Κάναμε αυτό το οποίο επιθυμούσατε να κάνουμε. Και έρχομαι εδώ στα σχόλια σε σχέση ε, με ε, τις ε, We had, um, as Commissioner, generally high compliance rate. σε σχέση με τα ποσοστά συμμόρφωσης των κοινοτικών υπηρεσιών. Φτάσαμε στο επίπεδο το 86% και άκουσα σήμερα την διαμεσολαβήτρια ότι το 15 θα φτάσει περίπου το ποσοστό συμμόρφωσης το 90% και θα πρέπει να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Εξετάζουμε φυσικά και το ποσοστό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί το 60% των υποθέσεων μας αφορά και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο έτσι ώστε να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο 100%. Ε, τα ποσοστά συμμόρφωσης ε, ε, είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει διαφορές ανατομέα, αλλά λαμβάνουμε σοβαρά τις παρατηρήσεις της διαμεσολαβήτριας και θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε όσο μπορούμε. Αναφέρθηκε και σε ένα θέμα στο οποίο δεν συμφωνήσαμε και θα επανέλθουμε στο θέμα της βιομηχανίας καπνικών προϊόντων αργότερα στα πλαίσια της συζήτησης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα κλείσω, Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας, ευχαριστώντας την εισηγήτρια ε, θα επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την εξαιρετική της συνεργασία με τη διαμεσολαβήτρια και τις υπηρεσίες. Και προσωπικά θα ήθελα να πω ότι η κυρία Οράιλη ε, πραγματικά της αξίζει ο τίτλος της υπερασπίστριας του λαού. Ε, ευχαριστώ. Περνάω τώρα στους ομιλητές. Το λόγο έχει ο κύριος Βαλέντσα. Δύο... Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την κυρία Ωράιλη για το έργο της, όχι μόνο για το 2014. Αλλά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της, η εργασία της είναι πραγματικά υποδειγματική. Η Επιτροπή Αναφορών στην έκθεσή της για τις δραστηριότητες της ε, διαμεσολαβήτριας περιλαμβάνει όχι μόνο σύνοψη του έργου της διαμεσολαβήτριας σε διάφορους τομείς, αλλά μας υπενθυμίζει κιόλας και σε θεσμικά όργανα ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ναι, ανοιχτή απέναντι στις προσδοκίες των πολιτών και στην ανύψωση του επίπεδου των διοικητικών υπηρεσιών. Η δυνατότητα, η εξουσία ίδιας πρωτοβουλίας για τη διενέργεια ερευνών της Ευρωπαίας Διαμεσολαβητίας μας δίνει και την απαραίτητη όθηση. Επ' αυτού θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στην προσπάθεια που καταβάλει η Διαμεσολαβήτρια για να επιτύχει μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς και για την στήριξη που δίνει στο Μητρό Διαφάνεια, το οποίο έχει δημιουργηθεί, ω γνωρίζετε, από κοινού μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανταποκριθούμε στι ανησυχίε του κοινού. Πάνω από 7.000 οργανώσει έχουν καταχωριστεί εθελοντικά. Και μόλις πριν από μία εβδομάδα άλλες 49 υπέγραψαν. Δείχνει αυτό μια εβδομαδα αλλε 49 υπεγραψαν δειχνει αυτο μια προθυμια για τη διασφάλιση της διαφάνειας που τη θεωρώ πολύ σημαντική πιστεύω ότι οι προφορίες που περιλαμβάνει το Μητρό για την αντιπροσωπευτικότητα των διαφόρων ε, μερών ε, πρέπει και αυτή να προωθηθεί και νομίζω ότι θα επιτρέψει σε εμάς εμάς που λαμβάνουμε αποφάσεις εν τέλει να γνωρίζουμε και να κατανοούμε καλύτερα τι πρέπει να πράξουμε ως Ευρωπαϊκή Θεσμή και ως Ευρωπαϊκή Ένωση το σύνολό της για να αντιμετωπίσουμε τα ε, προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μεσολαβήτρια. Ε, ευχαριστώ για ένα λεπτό τώρα. Η κυρία Μίτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από 23.000 πολίτες ζήτησαν την βοήθεια της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Μέγας αριθμός που δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει η Ευρωπαία Ombudswoman. Ο ρόλος της είναι σημαντικός για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα ε, των Ευρωπαίων πολιτών και να καταστεί πιο αποτελεσματικό το έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ώστε και οι πολίτες να βλέπουν με πιο ευνοϊκό μάτι το έργο των ευρωπαϊκών ε, θεσμών. Ωστόσο, να μην γελιόμαστε, χρειάζεται και άλλη δουλειά. Πολύ για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η χρηστή διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζεται και στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα. Η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να συμβάλλει ώστε να μπει ο πολίτης στην καρδιά των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την έκθεση της διαμεσολαβήτριας κυρίας Ορέιλη καθώς και βεβαίως και με την έκθεση της κυρίας Ρουίθ. Ο κύριος Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζουμε την εδώ παρουσία της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της κυρίας Οράιλη, και την συγχαίρουμε για την πανηγυρική επανεκλογή της. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 αναδεικνύει τη σημαντική δράση του οργάνου αυτού στη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, που αποτούν πλέον ενδυνάμωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο σε σχέση με τα θεσμικά της όργανα αλλά και με άτυπα όργανα όπως είναι το eurogroup και η τρόικα που λαμβάνουν ως γνωστό σκληρά και συνακόλουθα αντικοινωνικά μέτρα τα οποία επιβάλλουν στις χώρες που τέθηκαν σε μνημόνιο. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγκάστηκε μετά από ενέργειε τη διαμεσολαβήτρια να δημοσιοποιήσει την επιστολή τη προ την Ιρλανδική κυβέρνηση για την οικονομική κρίση. Οπότε και αποδείχθηκε πανηγυρικά η επεμβατική πολιτική της ΕΚΤ απέναντι στην Ιρλανδία. Όμω πρέπει να γίνουν ακόμα σημαντικά βήματα σε σχέση με τον έλεγχο τη λειτουργία τη Τρόικα. Γι' αυτό η διαμεσολαβήτρια οφείλει να διερευνήσει τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ω μέλο τη Τρόικα, ω πιστωτή των κρατών μελών του Μνημονίου και τη εντολή που έχει η ΕΚΤ με βάση τη συνθήκη. Το ίδιο ισχύει και για την σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο τη Επιτροπή μεταξύ του ρόλου που έχει η επιτροπή στην τρόικα και της ευθύνης της ως θεματοφύλακα των συνθήκων. σε μια φάση έντασης των προσφυγικών ροών πρέπει να υπάρχει έλεγχος και λογοδοσία της ίδιας της frontex ενώ σε σχέση με την ttip είναι δεδομένο ότι πρέπει η διαμεσολαβήτρια να εντείνει τη δράση της γιατί υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας. άλλωστε οι ευρωβουλευτές έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της TTIP μόνο με σκληρούς όρους εμπιστευτικότητας που παραβιάζει την δημοκρατική αρχή και εγκαθιδρύει καθεστώς μυστικής διπλωματίας. Μάλιστα μέχρι πρόσφατα οι υπουργοί των κρατών μελών της Ένωσης για να λάβουν τον έγγραφα της TTIP έπρεπε να πάνε να επισκεφτούν τις κατατόπους πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο της διαμεσολαβήτριας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά. Η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, κυρία Βίξτρομ, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με τη σειρά μου επιθυμώ να συγχαρώ την Έμιλι Ορέιλι, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, για την θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει. Αλλά και προσωπικά, Έμιλι, σας ευχαριστώ για την πολύ θετική συνεργασία μεταξύ ημών και του θεσμού σας και της δικής μου επιτροπής. Είναι πάντα πραγματική ευχαρίστηση η συνεργασία μαζί σας. Συνεχίζει στα ε, Σουηδικά η κυρία Βίξτρομ. Έλεγα λοιπόν ότι η διαμεσολαβήτρια ε, έχει επικεντρώσει την προσοχή της ιδίως σε θέματα διαφάνειας, διαφάνειας και ανοιχτής διακυβέρνησης που είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα για τον πολίτη. Στηρίζει έτσι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να γίνουν πιο ανοιχτά, πιο φιλικά στους πολίτες και πιο αποτελεσματικά, έτσι ώστε να κερδίσουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μιλούμε για το έτος 2014 και ένα από τα θέματα που ήταν πολύ σημαντικά τότε ήταν σχετικά με την Frontex, γιατί η Frontex πρέπει να λάβει επαρκές υλικό αλλά και προσωπικό, να έχει στη δηλαδή επαρκές υλικό και προσωπικό για να μπορεί να φυλάσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασπάζεται τις απόψεις της ε, Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και προτίθεται να δημιουργήσει μηχανισμό για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων καταγγελιών για παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Χαίρομαι επίσης που έχει προβλέψει και τη σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εγώ γνωρίζω βεβαίω καλύτερα από όλε τι άλλε χώρε την Σουηδία, την πατρίδα μου. Εκεί, σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπάρχει ακόμα πολύ άγνοια. Και αυτό είναι ανησυχητικό, διότι αυτό περιορίζει και την δυνατότητα των πολιτών να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Για μια στέρεα δημοκρατία είναι αναγκαίο οι αποφάσεις των πολιτών να βασίζονται σε γνώση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, είναι αναγκαίο ε, να συζητήσουμε όλες και όλοι πιο ενεργά με τους πολίτες να βελτιώσουμε τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι θεσμοί πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για τον διάλογο με τους πολίτες. Αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει και μπορούμε να συμβάλλουμε να έχουν μεγαλύτερη και βαθύτερη γνώση οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και πάλι προσωπικά την Έμιλι Ωραίλη. Σας ευχαριστώ. Αλμπιόλ Γκουσμάν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο στην έκθεση για την διαμεσολαβήτρια είναι η έλλειψη διαφάνεια στα ευρωπαϊκά όργανα και το πως οι θύρες που ανοίγουν ουσιαστικά πάντα για τα λόμπι κλείνουν ακριβώς εκεί που δεν πρέπει στο πρόσωπο των πολιτών. Ε, το πιο σοβαρό θέμα ήταν ε, οι διαπραγματεύσεις με το TTIP. Ε, δύο σημαντικές παρεμβάσεις της διαμεσολαβήτριας σε σχέση με τη μη δημοσίευση κάποιων εγγράφων ε, ταυτόχρονα σύμφωνα με αυτά παρά τις οδηγίες της διαμεσολαβήτριας αυτή η αντίληψη περί ε, κρυφής μυστικής λειτουργίας με τις πόρτες διπλοκλειδωμένες συνεχίζεται. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά μυστικά σε σχέση με αυτά τα οποία μας αφορούν και θα μετά από τα 3 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που υπέγραψαν κατά του TTIP εξακολουθούμε να μην έχουμε αποτέλεσμα. Η κυρία Άουκεν δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της και για το πνεύμα συνεργασίας. Να ευχαριστήσω και την Έμιλι Ρέιλι. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί αποδεικνύει συνεχώς ότι είχαμε δίκιο που την επιλέξαμε. Είναι μια πραγματική διαμεσολαβήτρια και όχι απλά μια προσωπικότητα καρπός μιας χαλαρής πολιτικής συνένεσης. Το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ε, να συνηθίσει ότι υπάρχει ένας σημαντικός διαμεσολαβικής. Θα συμφωνήσω με όλα αυτά τα οποία είπες Ευχαριστώ επίσης και για ό,τι έχεις κάνει για το Frontex και ό,τι σημαίνει αυτό για τη διαφάνεια. Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια και για το TTIP και για το Frontex. Πρέπει να συνεχίσεις την προσπάθεια επίσης και για την καλύτερη διαχείριση των ευρωπαϊκών οργάνων έτσι ώστε να εξυπηρετούνται πραγματικά οι πολίτες να δίδουν μια ξεκάθαρη και γρήγορη απάντηση να παίρνουν τις απαιτούμενες ε, συχνά εξηγήσει. Και αυτό θα πρέπει να διαπεράσει το σύνολο του συστήματος του Διοικητικού της Ένωσης, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Το θέμα της σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα πρόβλημα, δεν έπρεπε να υπάρχει, δυστυχώς όμως συνεχίζεται επειδή υπάρχει μια δήλωση για πιθανές ε, συγκρούσεις και επικαλύψεις συμφερόντων, αυτό δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν συμφέροντα και ουσιαστικά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει δεν είναι η ιδιωτική του ζωή, αλλά θέλουμε να μην υπάρχει ούτε κατελάχιστον σε επίπεδο επαγγελματικό μια σύγκρουση συμφερόντων. Και αυτό είναι το σημαντικό και έχουμε και προβλήματα επίσης και για την υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε προβλήματα στις δυνατότητες πρόσβασης στη δικαιοσύνη που δεν γίνεται σεβαστή σε διάφορες χώρες, αν και εδώ θα έπρεπε οι εθνικοί διαμεσολαβητές να ασχοληθούν περισσότερο. Έχεις το δικαίωμα να ερευνάς και στο Κοινοβούλιο, έχεις και υποχρεώσεις απέναντί μας και θα πρέπει να σεβαστείς και τις υποχρεώσεις αυτές. Ευχαριστώ κυρία Όκεν. μισή λεπτό. Ε, Εύη, πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την διαμεσολαβήτρια για την προσπάθεια την οποία έκανε. Ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική η παρέμβασή της έτσι ώστε να καταστούν πιο διαφανείς οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τα ευρωπαϊκά όργανα. Όπως είπαμε, οι περισσότερες καταγγελίες και έρευνες αφορούν την δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα, όπως επίσης και θέματα διαφάνειας. Πολλές φορές οι αιτήσει πρόσβασης δεν ικανοποιούνται. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ερευνηθεί ακόμα περισσότερο η διαφάνεια με την οποία διαχειριζόμαστε τα διαρθρωτικά ταμεία διαφορετικά ταμεία τα οποία σήμερα δεν είναι κάτω από ένα σοβαρό αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό. Επίσης, όπως δείχνουν οι εκ των υστέρων λογιστικές έρευνες, πολλές φορές υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε αυτούς που ελέγχουν και στους ελεγχομένους και πολλές φορές δεν αποδίδουν την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία προς ε, στους πολίτες. Σαν παράδειγμα το σχέδιο ΤΑΒ, ε, ταχεια συνδρομικη Σιδηρομική Σύνδεση Λιών-Τωρίνο. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους τοπικούς πληθυσμούς, εκφράζονται τα προβλήματα αυτά εδώ και χρόνια και όμως χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκές πιστώσεις. Πρέπει λοιπόν ε, και με τέτοια θέματα σε συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο να παρεμβαίνει η διαμεσολαβήτρια έτσι ώστε τέτοιου είδους ε, απαράδεκτες ε, προτάσεις να μην περιλαμβάνονται στις εργασίες μας. Ο κύριος Λεμπρετών, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση θέλει να δώσει απαλλαγή ε, στα πεπραγμένα της κυρίας Σορέλη για το 2014. Ξέρω ότι προσπάθησε να βελτιώσει τη διαφάνεια της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τομέα αυτό έλαβε δύο πρωτοβουλίες που πρέπει να ε, χαιρετήσουμε. Σε ό,τι αφορά τα λόμπις, ζήτησε και πέτυχε τη δημιουργία Μητρώου Διαφάνεια. Πάνω από 7.000 ομάδε πίσω έχουν εγγραφεί σε αυτό το Μητρό, το οποίο σίγουρα δεν θα επηρεάσει την επιρροή των 35.000 λομπιστών σε αποφάσει τη Ένωση, τουλάχιστον όμω υπάρχει και κάτι και αυτό. Κυρία Οράιλι, ε, πετύχατε επίσης να βελτιώσετε τη διαφάνεια και στις κλινικές δοκιμές. Οι πληροφορίες για τις κλινικές δοκιμές εν μέρη πλέον θα δημοσιεύονται και ιδίω ε, εκεί όπου γίνεται λόγος για την έγκριση κυκλοφορίας φαρμάκων στην αγορά. Οπότε θα μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερα για το βαθμό ε, της αποτελεσματικότητας ε, των φαρμάκων και του κώδικο των ερευνών. Βέβαια αποτύχατε να πετύχετε πραγματική διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις της Διατλαντικής Συμφωνίας TTIP. Σίγουρα κάπως έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά η διαβούλευση με τους ε, Ευρωβουλευτέ βουλευτές και όχι μόνο είναι προβληματική. Τελικά ε, παρακολύεται το πραγματικός ε, έλεγχος ε, αύριο, θα ακούσουμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν ε, δικαιούνται να ψηφίσουν αυτή τη συνθήκη που παρόλα αυτά θα δημιουργήσει κλειδονισμούς στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένα πολιτικό σφάλμα επίσης διαπράξεται κυρία Ράιλε ζητώντα να εφαρμοστεί η διαδικασία υποβολής καταγγελίας ενώπιον του Frontex από τους ατοντές άσυλο. Αυτή η διαδικασία πιστεύω θα χρησιμοποιηθεί από τους ε, μετανάστες για να παραμείνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλους αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσω την έκθεση. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει τώρα η κυρία Μορβάη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θαυμάσιο πρωινό πάλι εδώ στις Βρυξέλλες, ηλιόλου στο έξω, θαυμάσια ατμόσφαιρα εδώ στην αίθουσα ε, της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια θαυμάσια ατμόσφαιρα Πρόκειται βέβαια σήμερα για την ετήσια έκθεση της διαμεσολαβήτριας των ε, από τους 750 τόσους 25 βουλευτές ε, παρευρίσκονται σήμερα στην αίθουσα και συνομιλούν για το πώς θα γίνει πιο δημοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να την αγαπήσουν περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ιδίω βέβαια οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, γιατί αυτά τα θέματα σας απασχολούν σήμερα εδώ. Έχω μια ιδέα. Τι λέτε να ακούσουμε καλύτερα την φωνή των πολιτών, οι οποίοι λένε ότι ναι μεν νιώθουμε συμπόνια για τους ε, φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν ε, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους πολέμους που έχει ξεκινήσει η Δύση, αλλά εγώ σας λέω σταματήστε τις ροές των προσφύγων διότι επ' αυτού πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Και ανταυτού τι κάνετε. Ανέχεστε να καταπατούνται τα δικαιώματα των ανθρώπων που θέλουν ωστόσο, των Ευρωπαίων πολιτών, που θέλουν ωστόσο να υπερασπιστούν τις πατρίδες τους. Ενώ η αληθινή δημοκρατία είναι εκεί. Και αν χρειαστεί θα αγωνιστούμε κιόλας όπως κάνουμε εμείς στην Ουγγαρία που ε, θα διεξάγουμε δημοψήφισμα για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει δημοκρατία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρη, μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ε, διαμεσολαβήτρια κυρία Ορέιλι η οποία σε συνεργασία μάλλον η οποία η συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών είναι καλή. Είχαμε δώσει τρία αστέρια τότε στον προκάτοχό σα, τον καθηγητή Διαμαντούρο, για τη συνεργασία του μαζί μας. Θα μπορούσα να σα δώσω και ένα τέταρτο αστέρι σε εσά σήμερα. Εμείς επίση η πολιτική μου ομάδα θεωρεί δηλαδή ότι η έλλειψη διαφάνειας οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης. Η έλλειψη εμπιστοσύνης οδηγεί σε διάφορε φήμε και οι φήμε οδηγούν σε απώλεια αξιοπιστία. Διαφάνεια λοιπόν Όντως οι ε, ευρωβουλευτές έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και τους παρακαλώ μάλιστα και τους προσκαλώ να ε, ε, χρησιμοποιήσουν την πρόσβαση αυτή για να μην υπάρχουν τέτοια θέματα για την TTIP, για το Μητρό Διαφάνειας. Απόλυτη υποστήριξη εκ μέρους μου. Παρακαλώ μόνο στη συγκεκριμένη πλέον εφαρμογή να φροντίσετε η διαδικασία εφαρμογής να παραμείνει ε, λειτουργική. Ποιες επιφυλάξεις μπορεί να υπάρχουν. Χρειάζεται ταχύτερη προώθηση των καταγγελιών των πολιτών. Έχουμε βεβαίω την Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβήτρια, την Επιτροπή Αναφορών, έχουμε την Επιτροπή, μάλλον συγγνώμη, την Όλαφ, δηλαδή την Υπηρεσία των Σαπατών και ούτω καθεξής. Πρέπει να διοχετεύονται οι καταγγελίες στον σωστό αποδέκτη. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ λοιπόν για το έργο σα έω τώρα και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη έκθεσή σα. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Φρουντζουλίτσα. Μάλιστα, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Όπως γνωρίζετε, η διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε διάφορες έρευνες το 2014 και 2015 έχοντα υπόψη αυτή την ε, πάρα πολύ άσχημη κατάσταση με του ε, πρόσφυγε που διαιρεί τι ευρωπαϊκέ χώρε, δεν πιστεύετε ότι η διαμεσολαβήτρια θα έπρεπε να ξεκινήσει έρευνα για το πώ γίνεται σεβαστή από τα κράτη-μέλη η συμφωνία του χώρου Σέγγεν και πώ αυτό επηρεάζει του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Εσείς Πρώτη παρατήρηση. Είναι σωστό που εγκύπτει στο θέμα αυτό η διαμεσολαβήτρια. Και δεύτερο, για να είμαι ειλικρινής, όντως το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αυτό που ξέρω εγώ είναι μια οικογένεια πρέπει να είναι ενωμένη. Εγώ βλέπω οι διάφορε χώρε να φεύγουν προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό και υποστηρίζω απολύτως τη διαμεσολαβητία. Δεύτερο ή τρίτο, όλοι οι θεσμοί και το Κοινοβούλιο και η Διαμεσολαβήτρια και η Κομισιόν πρέπει να καθίσουμε κάτω να ψάξουμε να βρούμε μια λύση. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για περιγραφές των προβλημάτων, ενδιαφέρονται να υπάρξουν λύσεις προβλημάτων. Γι' αυτό χρειάζεται να εγκύψουμε όλοι με τόπο εντατικό στην προσπάθεια εξέβρεση μιας λύσης. Ένα λεπτό κύριε Γκυλιόμ. Είναι πολύ δύσκολο να αναφερθεί κανείς σε όλες τις δραστηριότητες της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας γιατί είναι πολλαπλές αλλά αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα που έχει απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα σταματήσω, θα σταθώ σε ένα θέμα στον τομέα της διαφάνειας στα πλαίσια του λόμπινγκ και των ευρωπαϊκών οργάνων. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων εφόσον θέλουμε να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό υπάρχουν και οι κώδικες δεοντολογίας να πω ότι οι προσπάθειες ξεκίνησαν όχι μόνο από εσά αλλά και από το 2011 και το θυμίζω αυτό στον συνάδελφο του Εθνικού Μετώπου που πήρε το λόγο προηγουμένως. Αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο δεν συμμετέχει στην προσπάθεια, δεν υπακούει στους ίδιους κανόνες. Το Συμβούλιο λοιπόν. Μήπως θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή όπως η Ανώτατη Αποπτική Αρχή για τη Διαφάνεια στην Πολιτική στη Γαλλία έτσι ώστε να ερευνάτε και να ανοιχνεύετε η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιθυμώ και εγώ κυρία Ορέιλη να σας ευχαριστήσω. Ο μέγας αριθμός ερωτήσεων προς εσάς και την ομάδα σας αλλά και η έκθεσή σας που ψηφίζουμε σήμερα δείχνουν πόσο καλό είναι το έργο σας για την βελτίωση της Ευρώπης κάτι που εγώ υποστηρίζω απολύτως για λογαριασμό της ομάδας μου, δηλαδή των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Είναι σημαντικό, ωστόσο, και αποδεικνύεται ότι σωστά εκλέξαμε μια γυναίκα με την πείρα σας από το εθνικό επίπεδο σε αυτή τη θέση. Για το θέμα TTIP, εάν ξεκινήσετε μια ίδια πρωτοβουλία για να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει τους κανόνες της διαφανείας. Πολύ σωστό. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για την προσπάθειά σας και για το έργο σας. Δίνετε μεγαλύτερη βαρύτητα και μεγαλύτερη ορατότητα, προσφέρετε, στην, ε, στον άγνωστο ακόμη για πολλούς θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κυρία Ρέιλι σας καλωσορίζουμε με ικανοποίηση στο Κοινοβούλιο για την Επιτροπή Αναφορών της οποίας ε, είμαι μέλος. Είστε το alter ego μας. Ε, είμαστε στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, έχουμε εργαστεί με συντονισμό με το δικό σας γραφείο. Υπάρχει αλληλεπίδραση και είναι πολύ ικανοποιητική συνεργασία κυρίως γιατί είστε αποφασισμένοι και γιατί μας δίνετε αποτελέσματα. Βελτιώνει ε, την διοίκηση η δράση σας ε, και η δέσμευσή σας μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό διότι με αυτές τις περιστραφόμενες πόρτες, ε, με το TTIP, με τις κλινικές δοκιμές με την επικοδομητική ματιά που ρίχνεται στο Frontex, ε, με το σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Όλα αυτά τη δείχνουν δουλειά, δείχνουν αποτελέσματα και αυτό εμπλουτίζει την κοινή μας δουλειά. Θέλω προσωπικά να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας στο μεταναστευτικό και το προσφυγικό, όχι για το 2014 μόνο, αλλά και το προηγούμενο έτος ε, που αναγκαστήκαμε να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Χρειάστηκε να δοθεί από την αρχή μια κοινή απάντηση. Είχαμε κάποιε συναντήσει κατά το παρελθόν και είχαμε συζητήσει τον ειδικό χαρακτήρα τη εντολή σα, του γραφείου σα. Ε, μια ψηλή απόδοση ομάδα που είναι στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, χαιρετίζω, επικροτώ τι προσπάθειέ σα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Και τώρα για ένα λεπτό το λόγο η κυρία Κούνεβα. Πιστεύόμαστε στην Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια γιατί παραμένει ένας από τους ελάχιστους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξίζει να, να εμπιστευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Την ώρα που η Ευρώπη βιώνει τη μεγαλύτερη υπαρξιακή της κρίση που οδηγεί αδυνατή να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως μαρτυρούν οι εικόνες των ταλαιπωρημένων προσφύγων, εικόνες που μας γυρίζουν στα δεκαετία του 30 ο θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι ένα στήριγμα διαφάνειας και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών. Επικροτούμε και στηρίζουμε την έκκληση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προς τη Frontex τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού ατομικών καταγγελιών για παραβιάσεις των τεμιλιώδων δικαιωμάτων των προσφύγων και την καλούμε να ερευνήσει περισσότερα το το ζήτημα στρέφοντας την προσοχή της στο δράμα που εξελίσσεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους Ευρωπαίους, στους ανθρώπους που εκπληρώνουν πίσω εκλυπαρούν πίσω από τα σύρματα και τα δικαιώματα στην ζωή και παραμένουν εκφοβισμένοι σήμερα στην Ιντομένη, στην Ατίνα και στον Περιά. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κύριο Σάρνοτ. Δεν είμαι εδώ για να ασκήσω κριτική στη διαμεσολαβήτρια που υπό δύσκολε συνθήκε κάνει μια δύσκολη δουλειά. 46% όμω των πολιτών δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα είναι πολύ ψηλότερο το ποσοστό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε υποθέσει για ανώτατου τραπεζίτες ε, και τι γίνεται όταν υπάρχει ε, κακή συμπεριφορά οι Beatles όταν τέλειωναν τις συναυλίες τους έλεγαν στο ακροατήριο είστε τόσο καταπληκτικό ακροατήριο θα θέλαμε να σας πάρουμε σπίτι μαζί μας αλλά δεν μπορούμε δυστυχώς πήραμε το προηγούμενο ακροατήριο και δεν χωράνε άλλοι. Θα μπορούσε αυτή να είναι Βρετανοί, Αν μπορούσαν να έρθουν εδώ στις Βρυξέλλες, να δουν τι βλέπουμε εμείς καθημερινά εδώ. Αν βλέπανε τις υπερβολές που γίνονται εδώ στις Βρυξέλλες ε, στις 23 Ιουνίου, σίγουρα θα ψήφισαν να φύγουν λεπτό. Εσταράς Φεραγκούτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τη διαμεσολαβήτρια Έμιλι Ρέιλι και για την επανεκλογή της και για την καταπληκτική της δουλειά. Ο τελικό στόχος ε, πάντα είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να παρέχουν ε, τις ε, βέλτιστες δυνατές δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες και βέβαια η εγγύηση των δικαιωμάτων των πολιτών είναι άλλο στόχος. Μιλήσατε για διαφάνεια, πράγματι ε, από τους στόχους και τις βασικές ε, διακηρύξεις ε, και θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο σας σε ό,τι αφορά τη νέα διαδικασία, τους νέους κανόνες για την επίτευξη του τελικού στόχου. Επίσης είστε συντονίστρα και για τις δικές σας πρωτοβουλίες. Εγώ θέλω να εστιάσω στην κακοδιαχείριση. Ένας από τους στόχους της διαμεσολαβήτριας είναι να έχουμε χρηστή ε, διαχείριση, χρηστή διακυβέρνηση. Τι θα πει αυτό, όταν ένα ε, δημόσιο οργανισμό δεν τηρεί ε, του κανόνε ή δεν τηρεί τι αρχέ τη Ένωση, μιλάμε για κακοδιαχείριση. Η οδηγία κατά των διακρίσεων που εδώ και έξι χρόνια έχει κολλήσει στο Συμβούλιο ή η μη επικύρωση της σύμβασης του Μαρακές για την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία αυτό δεν είναι κακοδιαχείριση. Ξέρω ότι είστε προσιλωμένοι ε, στην τήρηση της ε, σύμβασης για τα άτομα με αναπηρία. Σας παρακαλώ, ασκήστε την επιρροή σας στο Συμβούλιο για όσες χώρες ε, έχουν μπλοκάρει την οδηγία αυτή κατά των διακρίσεων και για τη σύμβαση του Μαρακές, γιατί μόνο έτσι θα τηρήσουμε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δύο λεπτά τώρα, κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Ρέιλε, ευχαριστώ και την ησυχήτριά μας. Η έκθεση υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που έχει να παίξει η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Είναι κομβικός ο ρόλος της έτσι ώστε να ακούγεται η φωνή του πολίτη. Ε, η κυρία Ράιλε έχει αποδείξει επανειλημμένα τον αγώνα τον οποίο δίδει για την διαφάνεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η έρευνα της διαμεσολαβήτριας για τις διαπραγματεύσεις TTIP που συνεχίζεται και σήμερα έχει μεγάλη σημασία για τον καθορισμό μιας σωστής εμπορικής πολιτικής. Επίσης διευκολύνθηκε η πρόσβαση σε εμπιστευτικά όγραφα θα πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι κάποιοι θεσμοί και όργανα όπως ε, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν βρίσκονται σε απειλή. Η Βρετανική κυβέρνηση θα μπορούσε πολλά να μάθει από σας κυρία Ωράιλη ε, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής της συμφωνίας TTIP στην λειτουργία του NHS, του, του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ υπάρχει σωστή συνεργασία ανάμεσα στη Διαμεσολαβήτρια και την Επιτροπή Αναφορών και είναι σωστή η πρόταση για την δημιουργία ενός κέντρου κατάθεσης παραπώνων για τους πρόσφυγες και μετανάστες των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από το Frontex όπως επίσης και οι κλινικές δοκιμές για τα φάρμακα είναι κάτι το οποίο όχι μόνο λειτουργεί προληπτικά σε επίπεδο διαφάνειας, αλλά θα βοηθήσει και τα ενδιάθεση στην αγορά φαρμάκων για την υπατήτη γάμα σαν παράδειγμα, με ευκολότερο και πιο ε, ασφαλή τρόπο. Πρέπει να συνεχίσετε λοιπόν την εφαρμογή του πενταετού σας προγράμματος και τη στρατηγική σας μέχρι το 2019 προς όφελος όλων μας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας και με την ομάδα σας. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Άρνοτ. Έχετε το λόγο κύριε Άρνοτ. Ευχαριστώ θέλετε εγγυήσει για το TIP ότι δεν θα επηρεάσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι διαφορετικό από αυτά τα οποία λέγουν οι, οι νομικοί εμπειρογνώμονες σε σχέση με τα λεγόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απορρίπτεται επίσης και τις συμβουλές τις οποίες έχουν δώσει τα Βρετανικά Συνδικάτα. Κοιτάξτε, παρανοήσατε εντελώς αυτό το οποίο είπα. Ε, πρέπει να υπάρχει δημόσια εμπιστοσύνη στις εμπορικές πολιτικές και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις νομικές συμβουλές ε, τις οποίες έχουν πάρει κάποια συνδικάτα όπως το Unite και όχι το Unison σε σχέση με τις επιπτώσεις μιας συμφωνίας για το TTIP στο δημόσιο σύστημα υγείας και τα συνδικάτα στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης και ε, διάφορες άλλες ομάδες ζητούν να δημοσιευθούν ε, οι απόψεις αυτές από πλευράς Βρετανικής κυβέρνησης. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της εργασίας της κυρίας Ορέιλη και η αφοσίωση στο έργο της είναι εγγύηση για το ότι θα ξαναδούμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας εκ μέρους της. Χαιρετίζω ιδίω την δέσμευσή της για την βελτίωση του έργου των ευρωπαϊκών θεσμών. Έχει σημειώσει τις παραλήψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων, κυρίως όσοι μιλούν για την ψηφιακή εποχή, πρέπει να αντιληφθούν ότι η ψηφιακή εποχή αλλάζει τα δεδομένα παντού και στην πολιτική. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από τη συνάδελφό σας. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία συνάδελφε, μιλήσατε για έλλειψη διαφάνειας και αναφερθήκατε στο παράδειγμα της TTIP. Μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση σχετικά με το πώς θα θέλατε εσείς να δείτε τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν σε διαδικασία. Αξιότιμη κυρία συνάδελφε, όσα διεξάγονται πίσω από κλειστές θύρες μπορούν να γίνουν και στο φως της δημοσιότητας. Οτιδήποτε άλλο δεν θα ικανοποιήσει τους ανθρώπους. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνονται αυτά με κλειστές πόρτες. Η κυρία Ιάτεν Μάκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου επιθυμώ να ευχαριστήσω την ε, διαμεσολευήτρια κυρία Ορέιλι για την θαυμάσια εργασία της. Επιθυμώ λέγω να την ευχαριστήσω την ίδια και το προσωπικό του γραφείου της για την πολύ αποτελεσματική εργασία της. Σύμφωνα με την έκθεση, το γραφείο της διαθέτει 67 συνεργάτες. Μα θα χρειαζόταν πολύ περισσότερους για να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό το έργο της. Παρ' όλα αυτά είναι αξιοθαύμαστο. Έχω ωστόσο μία επιθυμία. Στην συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεσπίσει νομοθεσία για τη χρηστή διοίκηση. Για την ώρα έχουμε μόνο δεοντολογικούς κανόνες. Γνωρίζω ότι γίνονται προσπάθειες, αλλά ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο, σε αυτούς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι αντίθετοι. Όμως, οι κανόνες για τη χρηστή διοίκηση είναι πολύ σημαντικοί για τους πολίτες. Όμως πρέπει να επιβάλλονται και στους αξιωματούχους για την ώρα οι πολίτες δεν μπορούν να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αυτό είναι άσχημο και για τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν υπάρχει δηλαδή σχετική νομοθετική ρύθμιση. Σας ευχαριστώ. η κυρία Νίριάντα. Καλωσορίζω την έκθεση της κυρίας Οράιλη και τη συγχαίρω για την εξαιρετική της δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτό το γραφείο, ιδίω ε, λαμβάνοντα υπόψη στις υποθέσεις, ε, παραδείγματο χάρη έρευνα για την κοινή αληφτική πολιτική για να υπάρχει διαφάνεια, πρόσβαση στα έγγραφα είχε αρνηθεί η Κομισιόν την πλήρη πρόσβαση, τώρα όμως υποχρεούται να είναι ε, διαφανής. Το ίδιο με τη συμφωνία TTIP. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχει την εξουσία η διαμεσολαβήτρια συγκεκριμένες ομάδες ε, να τις υποχρεώνουν να δίνουν απαντήσεις και για περιπτώσεις συγκρούσης, ε, συμφερόντων. Πρέπει να είναι διαφανής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρουμε πόσο δικαιολογημένα καχύποπτοι είναι οι πολίτε για την TTIP. Η ροϊκή δουλειά άσκησε για την ΕΚΤΑ η Έμιλιο Ράιλι και το ΕΚΤ χρειάστηκε ε, να δείξει την επιστολή στην Ιρλανδική ε, κυβέρνηση για την ε, τραπεζική κρίση. Εξαιρετική δουλειά και πάρα πολλά άλλα κάνει η Εμιλή Ράιλι. Είναι σαφές λοιπόν ότι το γραφείο της Ζαμεσολαβήτριας λειτουργεί όπως πρέπει και όλο και πιο δυνατό γίνεται στην υπηρεσία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό τώρα έχει το κυρία Βίνμπεργκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. προστασία των προσφύγων. Είναι μια αρχή που μπορεί να τύχει ευρεία ερμηνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι πρόσφυγες που έρχονται στα σύνορα της Ένωσης είναι όμως οικονομικοί μετανάστες. Πολύ λίγοι ζητούν το καθεστώς του πρόσφυγα για ανθρωπιστικούς λόγους. Άρα θα έπρεπε να επαναπροωθηθεί η πλειοψηφία αυτών και ίσως καταναγκαστικά κάποιες φορές Βέβαια, ε, πρέπει να δούμε από πλευρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αυτό παραβίαση ή όχι. Ε, δεν πιστεύω. Η δημιουργία τώρα από την διαμεσολαβήτρια ενό γραφείου παραπώνων ή καταγγελιών από ετούντε άσυλο πρόσφυγε που ζητούν να ε, εξεταστεί η υπόθεση του γιατί θεωρούν ότι έπεσαν θύμα κακή μεταχείρισης. Νομίζω ότι ε, απλά ε, θα λαδώσουμε πιο καλά τα γρανάζια ενό μηχανισμού που δεν δουλεύει καλά. Αντίθετα πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση για το πρόβλημα το μεταναστευτικό. Σφαίρ είναι ο επόμενος ομιλητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως κάθε χρόνο έρχεται η έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα λάβει τη μορφή ψηφίσματος. Το έργο σας είναι σημαντικό και αναμένουμε εξάλλου πολλά από εσά. Όμως δεν έχετε επαρκείς αρμοδιότητες για το έργο σας. Δέχεστε καταγγελίες μόνο εφόσον αυτές αναφέρονται σε κάποιο θεσμικό όργανο. Οι δεμή οι καταγγελίες αυτές προωθούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Εγώ έχω μάλιστα και προσωπικές εμπειρίες από ε, αυτήν την διαδικασία. Είχα υποβάλει καταγγελία για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με την εξαγορά της ε, Πάτρια και ωστόσο αυτή δεν έγινε δεκτή. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να διαμαρτυρηθώ. Μήπως πρέπει να θέσει κανείς το ερώτημα αν είναι καν χρήσιμο ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ίσως να τον χρειάζεται η Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να έχει επαρκείς αρμοδιότητες για να μπορεί να αντιδρά όταν συμβαίνουν προφανείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμανς. Η έκθεση την οποία έχουμε εδώ είναι μια καλή έκθεση. Και όχι μόνο αυτό, είναι μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει πολλές αλήθειες και δίνει πάρα πολλές πληροφορίες που περιγράφουν σωστά το τι έχει συμβεί. Η συνεργασία με την διαμεσολαβήτρια δεν περιορίζεται στη σημερινή συνάντηση. Επανειλημμένα έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν. Υπάρχει τακτική συνεργασία με την υπηρεσία της διαμεσολαβήτριας. Να επιμείνω στο θέμα του μητρώου διαφάνειας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιδέα. Ένα δεύτερο θέμα είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χθες δημοσιεύθηκε μια έκθεση και επί τη βάση αυτής της έκθεσης ε, βλέπουμε ότι έχει υπάρξει χειροτέρευση ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες. Λοιπόν, θα ήθελα τις καλύτερες ευχές μου να σας μεταφέρω και να πω ότι υποστηρίζω την έκθεσή σας. Ευχαριστώ η κυρία Σπινέλη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ την υπηρεσπίστρια των, του λαού, όπως λέει εμφατικά η, η κυρία Σπινέλη. Βλέπουμε ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Frontex, γιατί υπάρχουν από τη μία αυξημένες μεταναστευτικές ροές και από την άλλη μία χώρα μάλλον μια, ένα σύνολο χωρών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που κλείνει όλο και περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν ε, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να επιτρέψουμε στον ελεγχόμενο να ελέγχει τον ελέγχοντα και σε ποιο βαθμό μπορεί ε, η Frontex να διασφαλίσει την ευμάρεια γενικότερα των ε, μεταναστών και προσφύγων μπορούν να γίνονται τελικά δεκτές οι καταγγελίες ανώνυμες ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τι γίνεται στην περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι καταγγελίες αυτές. Τσάκι, 1,5 λεπτό. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω για μια ακόμη φορά την κυρία Ωραίλη θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και τις έρευνες της διαμεσολαβήτριας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να δούμε τελικά σε ποιο βαθμό υπάρχουν εγγυήσεις για το σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών και στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής. Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξυπηρετούνται τα, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσετε να ασχολείστε με αυτό και θα θέλαμε να δούμε τελικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και για την πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό το μέσο θα είναι χρήσιμο εφόσον είναι εύκολο τελικά, καταστήσει εύκολο για τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Η Ήτρια υπογραμμίζει βέβαια τα βασικά προβλήματα που είναι η διαφάνεια και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Από την άλλη δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις ε, εργασίες του Συμβουλίου από τη μία και στην κακή ε, οργάνωση και διαχείριση από την άλλη της Ευρωπαϊκής Διοίκησης. Θα πρέπει να δούμε και ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του διαμεσολαβητή και ποιοι όχι και να βελτιώσουμε την κατάσταση ε, δίνοντας την δυνατότητα να υπάρχει σωστή πληροφόρηση. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική πληρέστατη έκθεση και ε, ευχαριστώ και τον κύριο Τίμερμανς που αναγνώρισε ε, την προστέμενη αξία του Ισπανού ε, συνηγόρου του πολίτη, όπως είπε, υπερασπιστή του λαού. Το ίδιο κάνει και η κυρία Οράιλη. Μας ενδιαφέρει κυρίως ο εξυγχρονισμός, ο δυναμισμός με τον οποίο φέρει σε πέρα στο έργο της η διαμεσολαβήτρια, σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμμετοχή των πολιτών, πολιτών, πολιτική ανταγωνισμού, ε, εμπορίου. Είναι σημαντική τομή. Πρέπει να δείξετε, κυρία Οράιλη, ε, περισσότερη ε, ενεργητικότητα σε ζητήματα που απτονται και του τύπου. Και έχετε και κάποιες συστάσεις από την εισηγήτρια στο σημείο 22. Η επικοινωνιακή πολιτική πρέπει επίσης να βελτιωθεί. Δυστυχώς εμείς θέλουμε να γίνει και μια παιδαγωγική δουλειά περί αναγνώρισης των αποτελεσμάτων. Είπατε ότι οι χιλιάδες υπάλληλοι εργάζονται καταπληκτικά ε, παρότι υπάρχουν περιορισμοί και οικονομικοί και πολλές φορές ε, ε, η υγεία τους πλήττεται. Στη χώρα μου να πω επίσης ότι έχουμε πολλές καταγγελίες. Θα έπρεπε ίσως να έχετε καλύτερη συνεργασία με περιφερειακούς και εθνικούς συνηγόρους του πολίτες, ώστε να μην καταλήξουν σε εσάς ως έσχατο καταφύγιο οι πολίτες, ενώ υπάρχουν άλλες αρχές που θα μπορούσαν προηγουμένως να προσφύγουν. Ευχαριστώ. Κύριος Μπενίτο Θηλουάγα τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρώτα απ' όλα να τονίσουμε τη σημασία ε, της προσωπικότητας ε, της Ευρωπαϊκής ε, Δύο Μεσολαβητρίας. Πολύ σημαντική προσωπικότητα για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τις υπερβολές ε, της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και Νομοθεσίας. Ε, και στο θέμα των προσφύγων, που είναι τα βασικά θύματα των υπερβολών ε, της Frontex και των εξωτερικών τυχών που έχει ψώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θέλω να εστιάσω ε, σε αυτές τις περιστρεφόμενες πόρτες και να ευχαριστήσω την κυρία Ράιλ για τις προσπάθειες ε, που κάνει στον τομέα αυτό. Δυστυχώς ε, όμως δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε και την Κομισιόνα στις προσπάθειές της. Κάθε μέρα αντίθετα δείχνει ότι χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια. Δεν επιτρέπει προσβασή στις πληροφορίες και στα έγγραφα. Πόσοι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι που εγκαταλείπουν τη θέση, όπως λέει το άρθρο 16, ε, μας ε, ε, περνάνε αυτές τις περιστραφόμενες πόρτες και δεν ξέρουμε τι κάνουν. Πρέπει να πάψει να ισχύει αυτή η ανακύκλωση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα λόμπι, ε, γιατί ουσιαστικά οι λομπίστες ε, ε, πιάνουν τη δημοκρατία όμοιρο και τελικά αυτά τα οποία υποστηρίζονται είναι μόνο τα ε, συμφέροντα ιδιωτών και εταιριών. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία προσέλκυσης της προσοχή του Προέδρου. Γιάκοφ Τσίτς είναι ο πρώτος ομιλητής. ούτσινινο Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις εργασίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει, αλλά υπάρχουν πολλά τα οποία μένει ακόμα να γίνουν. Οι προσδοκίες των Ευρωβουλευτών, όπως βλέπετε, είναι ιδιαίτερα υψηλές για το σύνολο των ευρωπαϊκών οργάνων και κυρίως από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Την χάνεται λοιπόν της υποστήριξης σχεδόν όλων των πολιτικών ομάδων της, αυτού του Κοινοβουλίου έχετε την τεράστια, το τεράστιο ποσοστό της θετικής γνώμης ε, της ε, δημόσιας μάλλον κοινής γνώμης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη στους Ευρωπαίους πολίτες και στα πλαίσια του TTIP και στα πλαίσια της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Thank η κυρία Χάουταλα, αλλά δεν την βλέπω. Οπότε περνάμε στον κύριο Συναδινό. Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η προσπάθεια της κυρίας Οράιλη είναι αξιέπαινη, λαμβάνοντας υπόψη το σύντομο χρονικό διάστημα από την εκλογή της. Ο ρόλος της ως Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας να βοηθά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να καταστούν περισσότερο ανοιχτά, αποτελεσματικά και φιλικά προς τον πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση, είναι λίαν δύσκολος η ιδέα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να συνάδει με περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο των θεσμικών τη οργάνων. λαμβάνοντα υπόψη το ευρωβαρόμετρο του περασμένου μαΐου η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ένωση είναι μόλι 40 αντίθετα η έλλειψη αυτής αγγίζει το. 46. επιπρόσθετα υπάρχει ένα 20 των προτάσεων της διαμεσολαβήτρια με τις οποίες τα θεσμικά όργανα δεν έχουν συμμορφωθεί. υπάρχει πολλή δρόμος ακόμα σε τομεί όπω η διαφάνεια το κράτο δικαίου η δεοντολογία η καταπολέμηση της διαφθοράς η διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στο δημόσιο τομέα οι διαφάνειες κλινικέ κλινικές δοκιμές και κυρίως ο ανοιχτός χαρακτήρας της διαπραγματεύση για την ttip. προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζω την αύξηση του ετησίου προϋπολογισμού του γραφείου της ευρωπαίας διαμεσολαβήτριας αλλά θα επιθυμούσα και την εξέταση της νομικής δέσμευσης των υποδείξεων αυτής. ευχαριστώ. Thank Ο Η ύπαρξη ε, της δυνατότητας διαμεσολάβησης ε, και γενικότερα οι δραστηριότητές σας είναι μια καλή εγγύηση ενίσχυσης της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη οι παρεμβάσεις της διαμεσολαβήτριας ε, ξεκινούν από συγκεκριμένες αναφορές και παράπονα των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, νομίζω ότι ένας πραγματικός διαμεσολαβητής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει όμως να λειτουργεί και προληπτικά. Πρέπει να είναι σε θέση δηλαδή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ακόμα και αν δεν υπάρχουν αναφορές των πολιτών έτσι ώστε να υπάρξουν διορθώσεις σε ορισμένες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και των πολιτών. Σαν παράδειγμα η υιοθέτηση από πλευράς της Δανίας που επιτρέπει από πλευράς του κράτους την κατάσχεση των τιμαλφών των μεταναστών είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας οδηγήσει σε παρέμβαση διότι είναι ε, φρικτή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν και αυτό και το θέμα της διαφάνειας να είναι βασική πρωτοβουλία των δραστηριοτήτων σας. Ευχαριστώ. Κλείνουμε τον κατάλογο των ομιλητών και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Τίμερμανς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τεράστια πλειοψηφία των μελών που μίλησε σήμερα εκφράστηκε θετικά για τις εργασίες της διαμεσολαβήτριας και την έκθεση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ε, επιμείνουμε σε αυτό, θα περιοριστώ σε δύο θέματα το πρώτο θέμα έχει σχέση με την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων TTIP. Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη αυτού του σώματος να μας δώσει παράδειγματα από άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις όπου επικρατεί περισσότερη ε, διαφάνεια από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προκαλώ αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι όλα θα πρέπει να είναι δημόσια δεν υπάρχει καμία διεθνής διαπραγμάτευση όπου κάποια τμήματα της διαπραγμάτευσης ε, να μην αντιμετωπίζονται σε εμπιστευτικό επίπεδο και για διάφορους λόγους. Και η μέθοδος που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γνωρίζουν το περιεχόμενο των εγγράφων αλλά να μην το δημοσιοποιούν είναι ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε οι εκπρόσωποι του λαού να είναι ενήμεροι χωρίς να παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες της εμπιστευτικότητας. Το άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω και το οποίο έχει ήδη τεθεί από πολλούς από εσά Πρόεδρε, είναι το θέμα της διαφάνειας. Εμείς θα ξεκινήσουμε μια δημόσια διαβούλευση για τη διαφάνεια τον επόμενο μήνα, προετοιμάζοντας μια δήλωση, πρόταση, την οποία θα κάνουμε προς το Συμβούλιο, για ένα υποχρεωτικό μητρό διαφανείας, το οποίο είναι το επόμενο βήμα στο οποίο θέλουμε να περάσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εφαρμόσουν τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζουμε σήμερα εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω λοιπόν ότι όλοι εσείς που είστε υπέρ της διαφάνειας για μας, για την Επίτροπη, να επιδείξετε το ίδιο επίπεδο ζήλου σχετικά με τη διαφάνεια από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως ε, του Συμβουλίου. Λοιπόν, συμφωνώ με την παρουσίαση της κυρίας Οράιλη και θα πρέπει να συνεχίσουμε την αποκοινού προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Η κυρία Ωράιλη να κλείσει τη συζήτηση. Για μια στιγμή. Κυρία Μορβάη. κυρία Μορβάη. Ε, επειδή ακούμε διάφορες παρεμβάσεις, ε, ίσως είναι καλύτερα αν θέλετε να αφήσετε τους ε, βουλευτές να μιλήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και για τις παρεμβάσεις όλων σας. Μου δίνετε θάρρος. Με ενθαρρύνετε να εργαστώ ακόμα σκληρότερα. Δείξατε κάτι στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη αξία, διότι το έργο μου δεν μπορεί να γίνει σωστά και όπως πρέπει χωρίς τον την ενθουσιώδη υποστήριξη και των μελών του Κοινοβουλίου, το... την οποία ένιωσα σήμερα. Όπως είπε και ο κύριος Τίμερμανς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μεγαλύτερη ε, μερίδα από όσους μίλησαν τάχθηκε υπέρ των αποτελεσμάτων του έργου μας. Βεβαίως μιλείτε για τη διαφάνεια. Εσάς σας απασχολούν οι ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας. Και αυτό πάλι οι τοποθετήσεις σας αυτές με ενθαρρύνουν να εργαστώ ακόμα πιο σκληρά με τη δική σας στήριξη ώστε να καταστούν όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πιο διαφανή. Ένα άλλο θέμα το οποίο θίξατε συχνά ήταν η συμφωνία TTIP. Γνωρίζετε ότι έχω αρχίσει μια έρευνα για την διαφάνεια ε, στις διαπραγματεύσεις TTIP. Έθεσα το ερώτημα που έθεσε και ο Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς, δηλαδή ποιος είναι ο κατάλληλος χώρος για την εμπιστευτικότητα μέσα σε μια ε, διεθνή συμφωνία και ποια, πρέπει, ποια έγγραφα πρέπει να ανοίξουν. Πάντως ένας ομιλητής μίλησε, ε, μία ομιλήτρια μάλλον αναφέρθηκε στο ότι σήμερα βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή. Όντως οι νέοι ιδίω έχουν πολύ εντονότερες προσδοκίες σε ό,τι αφορά την διαφάνεια των πάντων. Θα συναντηθώ με την Επίτροπο Μάλστρομ την επομένη Δευτέρα και θα συζητήσω μαζί της ορισμένα από τα θέματα σχετικά με την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία TTIP είναι πολύ σημαντικό πάντως για μένα, εάν πρόκειται να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, να λάβω και τις σχετικές καταγγελίες. Άλλο θέμα που σα απασχόλησε είναι και η Frontex. Σα ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σα για την διαδικασία αντιμετώπιση των καταγγελιών. Θα τα κάνουμε αυτά στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των διατάξεων που αφορούν την Frontex και θα εγκύψουμε στο ε, μεταναστευτικό για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με συλλογικό τρόπο ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους, ευχαριστώ την εισηγήτρια, ευχαριστώ και σας κυρία Πρόεδρε και επαναλαμβάνω ευχαριστώ όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ενδιαφέρον που δείχνουν για το έργο του γραφείου μου. Ευχαριστώ κύριε Ράλη. Το τελευταίο λόγο θα έχει η εισηγήτρια κυρία Καμπεθόνου Ρουίθ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης ε, για το έργο τους, γιατί αυτή η έκθεση είναι ε, αποτέλεσμα κοινή προσπάθειας. Θέλω να ευχαριστήσω και την διαμεσολαβήτρια, γιατί και αυτή ε, συνεισέφερε στην έκθεση. Και θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε. Όλους θέλω να ευχαριστήσω. Μου μένει μια θετική γεύση, ένας θετικός απολογισμός. Ξεκινήσαμε μια, ένα ωραίο ταξίδι μαζί. Αυτό είναι η κατάληξη. Ε, πιστεύω ότι όλοι ε, έχουμε επίγνωση το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαυτή και η Επιτροπή Αναφορών Εγγυώνται τη συμμετοχή των πολιτών είναι θεσμοί κλειδιά, πρέπει να στηριχθούν από όλα τα θεσμικά όργανα γιατί πρέπει πραγματικά να βάλουμε τους πολίτες στο επίκεντρο και να συμμετέχουν και αυτοί στα κοινοτικά δρόμενα. Ε, τώρα, πρέπει να τονίσω ότι όλοι υποχρεούμαστε να περασπιζόμαστε και να εκπροσωπούμε τους πολίτες, ο καθένας στο αξίωμά του. Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και ιδίως ευχαριστώ την κυρία Οράλη.